Ach so, ja. Okay. So, dann stimme ich zunächst mal das Amendment 5. Ψηφίζουμε για την τροπολογία υπαριθμών 45, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται μετά 94 και 95. Όχι, πρώτα το 94. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 95. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Και πάλι το ΕΛΚ είναι ένας παραπάνω από όσους δικαιούνται. Τώρα είναι εντάξει. Έκλεισε η ψηφοφορία. 20 19, 25, 19 κατά, τέσσερις εποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1-2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Για τη 15. Έκλεισε ψηφοφορία. 39 υπέρ, 4 κατά. Ήταν σαφέ, αλλά ρώτησα και ζήτησα ηλεκτρονική επαλήθευση γιατί πολλοί δεν σήκωσαν το χέρι του. Εγκρίθηκε λοιπόν η 101 παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 107 παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 16 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 16 ψηφίζουμε παρακαλώ έκλεισε η ψηφοφορία 27 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται η 108 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 110. Σε δύο τμήματα ψηφίζουμε. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ για το πρώτο τμήμα, λέει ο πρόεδρος, έκλεισε η ψηφοφορία. 28 υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται. Τώρα για το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική 3-1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 3-2 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 4 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα, μισό λεπτό, στην 125, υπέρ παρακαλώ. Κατά, μισό λεπτό. 125 είναι λέει κάτω-κάτω. Ναι, είναι στην επόμενη σελίδα κάτω κάτω. Πάμε στην ε, τροπολογία 125. Στη σελίδα 4 είναι η τελευταία, η 125. Ξανά από την αρχή. Υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αναφέρεται σε μία ε, βουλευτή, πρόεδρος, μιλώντας, ε, απευθυνόμενη σε αυτήν προσωπικά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. 136 παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 139. Υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 161. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 29 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 8-1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8-2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 31 παρακαλώ υπέρ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 32. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 176 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε για την 176. έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστικη 8 8-3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αν θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. 30 υπέρ, 15 κατά, ένας αποχή, εγκρίνεται. Η τροπολογία υπεριθμών 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ή 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ. Για... Ε, ψηφίζουμε για την 185. Έκλεισε η ψηφοφορία. 28 υπέρ, 14 κατά, 4 αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές. Η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Η 186 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 187 με την προφορική τροπολογία Έχετε αντιρρήσεις κατά της ε, προφορικής τροπολογίας. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ παρακαλώ της 187 κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 187 με προφορική τροπολογία ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 24 υπέρ, 19 κατά, 2 εποχές εγκρίνεται. 188 ε, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνεται. Η 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 42 μέχρι την 192 μπορούμε να ψηφίσουμε όλες αυτές από κοινού αν δεν διαφωνεί κανείς υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη ομάδα 43 μέχρι 198 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική παλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε για τη 49. Έκλεισε ψηφορία. εγκρίνεται. Η συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η δέλτα συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά πάμε στην 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 64 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται ή 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία για την 68. Εγκρίθηκε. Η 69 με την προφορική τροπολογία. Ε, υπάρχει κάποιο που να διαφωνεί με την προφορική τροπολογία από τη βλέπω όχι κατόπιν τούτου ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Η 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, η 6 υπέρ, κατά, αποχές υποθέτω ότι εγκρίθηκε η 72 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίθηκε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 72 έκλεισε η ψηφοφορία 23 υπέρ, 22 κατά, τσίμα τσίμα η ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Η τροπολογία υπερθμών 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Για την 7. 26 υπέρ, 19 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 73. Υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η 77 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 9 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 9. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Η συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 81 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές κατά την άποψή μου απορρίφθηκε λέει ο πρόεδρος, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ για τη 12. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 30 υπέρ, 16 κατά, καμία αποχή, εγκρίθηκε με σαφήνεια. Τροπολογία υπερθμών 91 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος. 43 υπέρ, 3 κατά, καμία εποχή, εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους συνεισηγητές και όλους τους άλλους.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 για την τροπολογία του προϋπολογισμού. Έχετε μπροστά σας τον κατάλογο ψηφοφορίας και νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε ενσώματι, unblock, εκτός εάν κάποιος διαφωνεί. Από ό,τι βλέπω κανείς δεν διαφωνεί, κατόπιν τούτου, από ό,τι βλέπω συμφωνούν όλοι, ωραία. Λοιπόν, ψηφίζουμε σώματι από την 1 έως την 13. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ηλεκτρικά, ε, τέλος πάνω, έκανε λάθος πολύ, ηλεκτρονικά ήθελε να πει. Έκλεισε η ψηφοφορία. 41 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Ε, και εδώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή. Επόμενη ψηφοφορία ε, πρόκειται για τις διαδικασίες και πρακτικές όσον αφορά τις ακροάσεις των επιτρόπων. Εισηγητής είμαι εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Και Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία υπερτιμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο υπαριθμών 3 ε, προφορική τροπολογία, δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς, από ό,τι βλέπω όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 10. Ε, καταπίπτει αυτή και πάμε στην 11. 11 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 11. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 33 υπέρ, 7 κατά, σαφές το αποτέλεσμα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να το δω. Η τροπολογία υπερθυμών 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 19 παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική μορφή παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Τέσσερις υπέρ, ένας κατά, καμία εποχή. Ευχαριστώ <laughs> πάρα πολύ τον εισηγητή. Τον υποφαινόμενο δηλαδή. <laughs> Ερχόμαστε τώρα στην εφαρμογή της Λευκής ε, Βίβλου και ο εισηγητής έπρεπε να φύγει σύντομα αλλά θα επανέλθει. So, Πάμε τώρα στην συζήτηση για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του και για τις μεταφορές. Έχουμε τον Βιμ Καμπ μεταξύ μας και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα. Πριν ξεκινήσω να σας πω κάποιες παρατηρήσεις εισαγωγικά. Να τονίσω καταρχάς ότι στην έκθεση αυτή κάνουμε μια μεσοπρόθεσμη ανάλυση των αποτελεσμάτων της Λευκής Βίβλου του 2011. Δεν πρόκειται λοιπόν για, έναν, για μια αναθεώρηση, αλλά μια, για, για ένα τελικό απολογισμό, αλλά για έναν ενδιάμεσο, προσωρινό. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε κατά πόσον οι προτάσεις εκείνες που είχαμε ετοιμάσει το 11 ε, ο κύριος Γκρός ήταν ο εισηγητής τότε ο προκατοχός μου και να εξετάσουμε κατά πόσον υλοποιήθηκαν οι προτάσεις. Να σας πω τα εξής. Το είπε και η κυρία Μπιλμπάου νωρίτερα τα κράτη-μέλη, το τονίζω αυτό, είναι πολύ πίσω στο χρονοδιάγραμμα. Έχουν καθυστερήσει πολλά ζητήματα. Για παράδειγμα, στις αερομεταφορές, αλλά και στα μέτρα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ως εκ τούτου. Αυτό που επήγει κυρίως πρωτίστως είναι να δώσουμε έμφαση στην πολιτική των μεταφορών. Άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Δεν θα ήθελα να κατηγορήσω κάποιο κράτος μέλος στην Ευρώπη. Όλα πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα που εγκρίθηκαν, αλλά πρέπει να τα εφαρμόσουν πολύ ταχύτερα, ε, με μεγαλύτερη έμφαση. Επίσης, πρέπει να επιλέξουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση στον ενδιάμεσο αυτό απολογισμό. Πρόκειται για μια φωτογραφία της κατάστασης. Δεν θέλουμε να ανατρέψουμε το πλαίσιο, θέλουμε μια συνέχεια ε, η οποία θα προχωρήσει και μετά την φετινή χρονιά. Να τονίσω επίσης την μεγάλη σπουδαιότητα του κλάδου των μεταφορών στην Ολλανδία λέμε χωρίς μεταφορές δεν κινείται τίποτα. Υπάρχουν κοινοβουλευτικές επιτροπές ωστόσο που πιστεύουν ότι το κοινοβούλιο, μιλώ για την ε, συνταγματική επιτροπή, την οικονομική επιτροπή που πιστεύουν ότι πρέπει να ασχολεί το κοινοβούλιο με άλλα θέματα, αλλά όλα τα θέματα που θέλουμε να ε, περάσουμε στην Ευρώπη δεν μπορούν να υλοποιηθούν αν δεν υπάρχουν μεταφορές. Η αλλαγή το, του τρόπου επικοινωνίας, αυτό το modal shift που λένε στα αγγλικά, δεν έχει επιτευχθεί, ίσως γιατί το θεσμικό πλαίσιο που επιβλήθηκε ήταν υπερβολικά ρηξικέλευθο, υπερβολικά απαιτητικό. Δεν άλλαξαν, δεν άλλαξε ο ανατολισμός των μεταφορών ωστόσο από τον ένα κλάδο στον άλλο. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε προς μια πολυτροπικότητα ή μια συντροπικότητα του κλάδου των μεταφορών, ούτω ώστε να μπορέσουμε να παροτρύνουμε αυτή την αλλαγή παραδείγματος στον χώρο των μεταφορών. Χωρίς να επιβαρύνουμε, χωρίς να, ε, να δημιουργήσουμε προβλήματα στις οδικές μεταφορές, απλά δίνοντας ε, έμφαση στην διεύρυνση των υποδομών, άλλων μέσων μεταφοράς, των σιδεροδρομικών γραμμών για παράδειγμα, της ποτάμιας μεταφοράς. Για το λόγο αυτό πρέπει να εμείνουμε στην ανάγκη να υλοποιηθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα, να επενδύσουμε όλο και περισσότερο στις σιδεροδρομικές μεταφορές, στις ποτάμιες μεταφορές, στόχους που είναι στόχοι βιώσιμοι. Βλέπουμε ωστόσο ότι η βιωσιμότητα δεν επιτυγχάνεται στον κλάδο των μεταφορών. Έγιναν πάμπολες προσπάθειες, υιοθετήθηκαν πολλά μέτρα, αλλαγή κινητήρων. Ωστόσο, οι στόχοι που τέθηκαν μέχρι σήμερα, που τέθηκαν το 2011, δεν επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει αναθεώρηση των στόχων βιωσιμότητας, αλλά θα ήταν σκόπιμο να γίνει προσπάθεια για να τους υλοποιήσουμε. Κάτι άλλο σημαντικό θέμα είναι το θέμα των αστικών μεταφορών που θα διπλασιαστεί. Εγώ αν προσπαθήσετε να έρθετε μια μέρα που βρέχει στο κοινοβούλιο και θα δείτε ότι η πόλη παραλύει. Ε, τα πάντα είναι μπλοκαρισμένα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις αστικές μεταφορές. Ξέρετε ότι εγώ προτιμώ τα ηλεκτρικά ποδήλατα εγώ θα ήθελα περισσότερες, περισσότερα τέτοια ποδήλατα στην πόλη. Τώρα, τα συστήματα έξυπνων μεταφορών θα βελτιώνει την κατάσταση, αλλά μπορεί να βελτιωθεί πολύ σημαντικότερα. Για παράδειγμα, χθε. εξετάσαμε την έκθεση του κυρίου Κόχ για την ενοποίηση των ε, εισιτηρίων. Υπάρχουν ωστόσο πολλά ε, τεχνολογικά εμπόδια τα διόδια, για παράδειγμα, τα συστήματα διοδίων, πριν προχωρήσουμε στην ενοποίηση του, των, της ηλεκτρονικής μεταφοράς πόρτα-πόρτα. Τα θέματα της, ε, των τελωνιακών ε, εντύπων που απαιτούνται για τις μεταφορές, των εντύπων που συνοδεύουν τις μεταφορές ε, εμπορευμάτων και αυτά πρέπει να ενοποιηθούν και να, γίνουν, να αποκτήσουν ηλεκτρονική μορφή. Τώρα, για την εσωτερική αγορά στην Ευρώπη, όταν μιλάμε για το, τις, τις επιπτώσεις, τις κοινωνικές επιπτώσεις των μεταφορών, οι οδηγοί αυτοκινήτων ε, φορτηγών στη Γερμανία, για παράδειγμα, που έχουν μια νομικά στέρεη θέση, η οποία ωστόσο υπονομεύεται στη Γερμανία και αλλού από τις εξελίξεις. Έχουμε και τους φίλους από το Uber που δημιουργεί νέα ζητήματα. Η πρόκληση του Uber είναι μια σημαντική ε, αλλά Εμείς είμαστε υπέρ του εξυγχρονισμού των μεταφορών, αλλά δεν μ' αρέσουν οι κοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο, να αποφεύγεται δηλαδή κάθε μορφή κοινωνικών, κοινωνικής προστασίας. Εμείς είμαστε υπέρ μιας κοινωνικής οικονομίας αγοράς. Δεν θέλουμε ένα καθαρά καπιταλιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Ε, άλλο θέμα. Η καθημερινή ασφάλεια. Ο κύριος Κόχ είναι ο μόνιμος εισηγητής ε, ακόμα, αλλά έχουμε ε, αύξηση των θυμάτων. 25.000 ε, νεκροί στους αυτοκινητόδρομους είχαμε το 2014. Η έμφαση τώρα δίνεται στην τρομοκρατία και τις εξωτερικές απειλές. Αλλά τι γίνεται με την σφαγή στους δρόμους μας. Και δεν μιλώ μόνο για τα θανατηφόρα ατυχήματα, αλλά και για τον τεράστιο αριθμό των τραυματιών. Το θέμα δεν είναι μόνο της ανθρώπινης οδύνης που είναι φοβερό, αλλά και όλες οι επιπτώσεις, ασφάλειες, ε, αναπηρίες, απόλυτα εισοδήματος, απώλεια εργατικού δυναμικού. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Αυτά ήθελα να σας πω εξ αρχής παρουσιάζοντας την έκθεση. Ευχαριστώ όλους σας, ιδίως τη Γραμματεία, για τη δουλειά που κάναμε. Πετύχαμε πολλά πράγματα. Είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω τις απόψεις, σχόλια και προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα η Κλάουντια Καπαντέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς να πω μάλλον συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που πέρασαν που έκαναν καθολικό Πάσχα, να χαιρετήσω και τους Ορθόδοξους συναδέλφους που είχαν Πάσχα προχθές. Μια σειρά παρατηρήσεων καταρχάς. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις παρατηρήσεις του. Είναι σαφές ότι η πρόταση αυτή ξεκινά από μια εξαιρετική αφετηρία, δηλαδή την υλοποίηση της Λευκής Βίβλου του 2011. Αυτό είναι αφετηρία για μας. Εγώ έχω προτείνει ως συντονίστρια των σοσιαλιστών μια σειρά τροπολογιών για να πετύχουμε ε, πολλές από τις παρατηρήσεις που παρουσίασε ο κ. Κάμπ. Μιλώ καταρχάς για την κοινωνική διάσταση. Είναι γεγονός ότι υπήρξε πρόοδος, ότι υιοθετήθηκαν ε, νομοθετικά κείμενα σε κάποιους κλάδους. Χρειάζεται ωστόσο μεγαλύτερη προσπάθεια για την εναρμόνιση της εργατικής νομοθεσίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να κάνει προτάσεις ούτως ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο εναρμόνισης των εργασιακών δικαιωμάτων ίσως με έναν οργανισμό ο οποίος θα εποπτεύει την εφαρμογή της ε, συγκεκριμένης νομοθεσίες, μια υπηρεσία ενδεχομένως για τις χερσέ μεταφορές. Εμείς δουλεύουμε με συναδέλφους από τους σοσιαλιστές για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων ε, το 2011, από το 2011 μέχρι τώρα εγκρίθηκαν κάποια νομοθετικά κείμενα. Θα ήθελα η έκθεση να παραπέμπει σε κάποια από αυτά τα στοιχεία. Για παράδειγμα, το πακέτο του 2013 για το κλίμα και την ενέργεια, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση, για παράδειγμα. Εμείς κάνουμε ένα εγχείρημα προσπαθώντας να υλοποιήσουμε στην πράξη τη Λευκή Βίβλο του 11. Για το λόγο αυτό, αυτή, αυτό το εγχείρημα είναι αναγκαίο γιατί πρέπει να αλλάξουμε ριζικά τον κλάδο των μεταφορών, ιδίω ε, είχαμε ε, μετά τις αποφάσεις του 2010. Αυτό ωστόσο πρέπει να γίνει με μια σφαιρική οπτική, αναγνωρίζοντας τις συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ του κλάδου των μεταφορών αφενός και της ενέργειας αφετέρου. Πρέπει να υποβάλουμε μια σειρά συστάσεων και σε άλλα ζητήματα όπως την ε, πολυτροφική έκδοση εισιτηρίων, την αστική οικολογική κινητικότητα. Οι συστάσεις των δύο ε, εκθέσεων πρέπει να υιοθετηθούν στις εργασίες μας. Τώρα, η βελτίωση της κινητικότητας της πόλης πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Άλλη, ε, μια άλλη τροπολογία μας αφορά τις διάφορες κατηγορίες πολυτροπικής μετακίνησης και την χρήση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των μεταφορών και της ασφάλειας της πόλης. Κάτι ακόμα, η αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την άνεση των επιβατών και την μετακίνηση. Τέλος, να επενδύσουμε τις υποδομές και να αυξήσουμε τις επενδύσεις στον τομέα αυτό. Το σύστημα των μεταφορών απαιτεί μια δυναμική ε, αλληλουχία των, ε, ε, υποδομών. Πρέπει να δώσουμε έμφαση σε καθαρές ε, υποδομές, σκεπτόμενοι και την ανάγκη των χωρών, τις ανάγκες των χωρών συνοχής. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί για τις τελευταίες αυτές χώρες η έμφαση στην, στις καθαρές υποδομές. Ε, δεν μειώσαμε ωστόσο ούτε καν τον αριθμό των θυμάτων ε, σε τροχέα. Ε, με άλλα λόγια, πρέπει να ελέγξουμε πώς εφαρμόζεται η Λευκή Βίβλος, να δούμε αν οι στόχοι επιτεύχθηκαν και να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο σύστημα έξυπνων και ασφαλών μεταφορών, εκμεταλλευόμενοι όλα τα υφιστάμενα κείμενα όχι μόνο τα επίσημα αλλά και όλες τις άλλες ιδέες που έχουν υποβληθεί. Ευχαριστώ. Θα υποβάλουμε τροπολογίες με του συναδέλφου Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Κόσμας Λοτόφσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κύριο Βιμ Βαντενκάμπ για την πολύ καλή του δουλειά και γιατί μας ε, παρουσίασε τα αποτελέσματα της δουλειάς του σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πολύ αποτελεσματικά, κάνει έναν απολογισμό των ζητημάτων και με πολύ συνοπτικό τρόπο, κάτι ασυνήθιστο στο σώμα, μας παρουσίασε τις προτάσεις του. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτές τις βασικές προτεραιότητες Πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι μοναδική η Ευρώπη, δεν είναι ωστόσο αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Σε όλε τις δράσεις λοιπόν που αναλαμβάνουμε να φέρουμε σε πέρας θα πρέπει να εντάξουμε τις ε, γενικότερες σε ένα γενικότερο ευρύτερο πλαίσιο να λάβουμε υπόψη μα. Ένα πολύ καλό παράδειγμα εδώ θα ήταν να ακολουθήσουμε ένα πιο αισιόδοξο χρονοδιάγραμμα ε, για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Μικρότερη εξάρτηση από τον άνθρακα και επειδή είναι χαμηλότερε οι τιμέ του πετρελαίου βλέπουμε ότι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε και την ανάπτυξη. Βλέπουμε τις προσπάθειε που γίνονται σε άλλε χώρες του κόσμου. Όταν όμως δεν μειώνουμε αυτή την εξάρτηση, μειώνουμε τις προοπτικές ανάπτυξης, τις θέσεις εργασίας κτλ. Επίσης, ελεύθερος ανταγωνισμός στον τομέα των μεταφορών. Πάλι πρέπει να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Τι κάνουν οι άλλες χώρες. Τι κάνουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Αεροπορικές εταιρείες, να σας δώσω ένα παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι λόγο των κεφαλαίων που επενδύουν οι αραβικές εταιρείες κερδίζουν το πνεύμα ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Αν παραμείνουμε παθητικοί ή μείνουμε σε κοινωνικά επιχειρήματα, θα γίνουμε και εμείς όλο και πιο προστατευτική. Και δεν θα μπορούν κάποιες ε, εταιρείε ε, ορισμένων κρατών μελών να ανταγωνιστούν με εταιρείε άλλων κρατών μελών. Και αυτό θα αυξήσει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Άρα δεν θα πετύχουμε τους στόχους του εγγράφου. Πιστεύω ότι θα πρέπει σίγουρα να εστιάσουμε στον άνθρωπο, στον επιβάτη, γιατί οι επιβάτες, οι καταναλωτές είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ωφεληθούν και από τις ε, φθηνότερες τιμές εισιτηρίων. Οι οδηγοί, οι ποδηλάτες επίσης θα πρέπει να είναι αυτοί που θα ευνοηθούν από μια νέα κουλτούρα ασφάλισης μεταφορές. Ωστόσο, μεταφορές σημαίνει και άλλα άτομα, παραδείγματος χάρη αυτοί που εργάζονται σε διελιστήρια πετρελαίου ή σε αυτοκινητοβιομηχανίες για αυτούς τους ανθρώπους, αν οι αλλαγές ε, γίνουν πάρα πολύ γρήγορα και αν υπάρχουν έντονες πιέσεις για απαλλαγή από τον άνθρακα, θα υπάρξουν απόλυες. Ας δούμε τι έγινε στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Οι διατροπικές μεταφορές, ώστε να μην είναι για αυτούς τους ανθρώπους ο βασικός στόχος. Ο βασικός στόχος θα ήταν η πρόσβαση στις μεταφορές. Πολύ πιο απλά. Θα πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν και στα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών των πολιτών. Ελπίζω με τι τροπολογίε να ληφθούν υπόψη και τα δικά μου επιχειρήματα τα οποία μόλι σα εξέθεσα. Είναι πολύ σημαντικό για την πολιτική μεταφορών των προσεχών ετών. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η Γκεστίνε Μάσινα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Βιφαντεκάμ, τον εισηγητή μας, ο οποίος είπε ότι επιθυμεί να έχει μια συμπυκνωμένη και εμπεριστατωμένη έκθεση και όχι αερολογίες. Και νομίζω ότι τα κατάφερε πάρα πολύ καλά γιατί η έκθεση είναι ισόρροπη. Ε, συναντήθηκε με τους σκιώδης ηγητές, με εμά δηλαδή, και ο καθένας μπορούσε να εκφράσει την ε, άποψή του και πράγματι αυτά που είπαμε τα έλαβε υπόψη σου. Παρόλα αυτά έχω και κάποιες παρατηρήσεις, όχι μόνο επένους, Λοιπόν, γράφεις ο ε, ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει modal shift και πολυτροπικότητα και τα δύο πρέπει να υπάρχουν, το να μετακινηθεί λιγάκι το πρότυπο, αυτό είναι σωστό, αλλά δεν φτάνει και το έχω πει αυτό επανειλημμένα, ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να μετακινηθεί η κίνηση από τους δρόμους ε, στη θάλασσα ή ε, σε άλλα μέσα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γίνεται λόγος για την πολυτροπικότητα. Επίσης γίνεται λόγος ε, για τις ε, υποδομές, γίνεται λόγος για ευθύ μεταφορικά συστήματα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στο χρήστη των μεταφορών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω αφορά την ασφάλεια των οδικών μεταφορών. Εκεί λοιπόν γίνεται παραπομπή στις καινοτόμες τεχνολογίες σε κυρίως όσον αφορά τα γιοταχή. Και θέλω να σας πω ότι επ' αυτού θα κάνω μία παρατήρηση, γιατί για μένα πολύ ωραία είναι όλα αυτά που μπορούν να προκύψουν ως καινοτομία και στα γιοταχή και στα φορτηγά, αλλά όλα αυτά έχουν σχέση με τη ροή δεδομένων. Θεωρώ λοιπόν ότι η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας ε, και των δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Ε, ξέρουν πάρα πολύ ότι εγώ έχω αγωνιστεί για την προστασία των ε, δεδομένων έτσι ώστε ε, να υπάρχει κάποια προστασία ακόμα και στο e-call, σε αυτό το αυτόματο σύστημα ζήτησης ε, ανάκλησης βοήθειας. Ε, θέλω λοιπόν να κάνω μία παρατήρηση. Ε, στον τομέα αυτό να υπάρξουν θέσει εργασία και για γυναίκες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές που θα ενδιαφέρονταν. Ίσως λοιπόν πρέπει να προσφερθούν κάποια κίνητρα. Κατά τα άλλα, οι μεταφορές ε, χωρίς χρήση χαρτιού και αυτό αναφέρεται και είναι πολύ σημαντικό ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τη ρήπανση γίνεται λόγος για το Παρίσι για την επικείμενη συνάντηση όπου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερη προστασία του κλίματος Κατά τα άλλα, όσον αφορά τους μεμονωμένους τομείς μεταφορών, θέλω να πω ότι στις αεροπορικές μεταφορές λείπει κάτι, δηλαδή η εσωτερική στρέβλωση ανταγωνισμού που υπάρχει και δεν αναφέρεται αναφέρεται. Και θέλω να πω το εξή. Υπάρχουν πολλοί που ακολουθούν το δικό του δρόμο, κάθε κράτο το δικό του. Όπω η φορολόγηση των επιβατών στην Αυστρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αν θέλετε υπάρχει το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί και να διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Γιατί όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των αερομεταφορών. Όσον αφορά τις σε οδικές μεταφορές. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να μιλάμε ήδη τώρα για ε, δεσμευτικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, κυρίως όσον αφορά τα φορτηγά, γιατί αυτά διαφέρουν ακόμα και όσον αφορά τις εκπομπές τους. Εξαρτάται από τα είναι μικρά, τα φορτηγά αν είναι μεγάλα. Εδώ εντάσσονται και τα λεωφορεία. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Εξ όσων γνωρίζω λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τη βιομηχανία προσπαθούν να βρουν ένα σύστημα πώ θα μετρώνται όλα αυτά και θα κατηγοριοποιούνται και μετά να γίνεται κάποιος έλεγχος. Κατά την άποψή μου να απαραίτητο να υπάρχει προκατακτική εργασία, να περιμένουμε και μετά ε, να ε, ορίσουμε δεσμευτικές ε, οριακές τιμές. Πολύ πιο καλό αυτό από το να προχωρήσουμε τώρα σε μία ρύθμιση ή σε έναν κανονισμό. Κατά τα άλλα υπάρχει και μία άλλη ρύθμιση για πάλι την πολυτροπικότητα που είναι πολύ σημαντική και για λογιστικά θέματα. Νομίζω ότι μπορούν να συνδεθούν πολύ καλύτερα μεταξύ τους ε, τα ηλεκτρονικά μηχανογραφικά συστήματα πάντα σε θέματα επιμελητίας και υποδομών. Ε, να μην υπάρχουν μόνο αερολογίες ε, ο μιλητής μίλησε πολύ για την αρχή ο, ο χρήστης πληρώνει, με βάση την αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει, αλλά δεν λέγεται τίποτα για το earmarking στις ε, υποδομές. Χρήματα τα οποία ε, εισπράττουμε από τις μεταφορές να τα επενδύουμε και πάλι στις υποδομές. Αυτές είναι οι βασικές μου παρατηρήσεις. Ε, σε πάρα πολλά συμφωνώ και εγώ ότι επιθυμούμε όλοι τον ενιαίο αεροπορικό χώρο. Θέλουμε ε, να υπάρχει ε, και ένα είδος σύμπνοιας ε, στην ναυτιλία. Έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, αλλά είμαι ευχαριστημένη με το σχέδιο. Πριν δώσω το λόγο στους επόμενους, θα ήθελα να καλωσορίσω μία ομάδα επισκεπτών. Ο κύριος Λάιχτφριτ κάλεσε μία ομάδα μία, της νεολαίας των σοσιαλδημοκρατών. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή μας. Spontan in der Debatte geht jetzt weiter mit Merja Kielön. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin... Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Κίλωνεν, καταρχάς να δώσω ε, συγχαρητήρια στον Βίμ για την πολύ καλή δουλειά του. Σε ευχαριστώ Βίμ. Και να πω ότι πράγματι υπάρχουν στην έκθεση στοιχεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να τροφοδοτήσουμε τον ευρύτερο προβληματισμό για αυτά τα θέματα. Θα μπορούσα να γίνει να πω ότι η Λευκή Βίβλος του 2011 έθετε πολύ ενδιαφέροντες στόχους, όμως δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη. Ως νομοθέτες έχουμε μία υποχρέωση. Πρέπει να θέτουμε στόχους περιβαλλοντικούς που να είναι υψηλοί, αλλά έχει σημασία και η ψηφιοποίηση. Πρέπει να πατήσουμε τον γκάζι, αν θέλετε τώρα, για να υλοποιήσουμε ό,τι αποφασίστηκε το 2011. Γι' Και αυτό θα ήταν καλό για να έχει η Ευρώπη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Επίση, δεν πρέπει να μα διαφεύγει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον παγκόσμιο ανταγωνισμό όλο και νέα πρότυπα, όλο και νέοι κανόνε, ε, νέα συστήματα πλοήγηση κτλ. που βλέπει το φω τη ημέρα. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό Δυστυχώς όμως εμείς στην Ευρώπη είμαστε ουραγοί. Παναπαυόμαστε στις δάφνες μας θα έλεγα. Και κλείνουμε και λίγο τα μάτια σε αυτή την ψηφιακή επανάσταση. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες για νέες υπηρεσίες. Με στόχο τους πολίτες, τους χρήστες, τους επιβάτες. Νέες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τους νέους τρόπους μεταφοράς. Επομένως, ζήτηση υπάρχει. Η προσφορά είναι αυτό που λείπει. Πιστεύω ότι αυτό που λείπει είναι να δεσμευθούμε περισσότερο στον τομέα των μεταφορών στην καινοτομία, στην εφαρμογή της καινοτομίας στην πράξη. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως, θα πρέπει να δώσουμε, να αφήσουμε χώρο για αυτές τις καινοτομίες, για να τις εκμεταλλευτούμε. Να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν νέες δυνατότητες με τα νέα συστήματα. Και οι καινοτομίες αυτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση να βρουν το χώρο τους, παραλαμβάνω. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα πρέπει να υποβαθμίσουμε τα πρότυπα ασφαλείας, τα περιβαλλοντικά πρότυπα ή την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Γιατί και αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Αν καταφέρουμε να εγγυηθούμε την ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των πτυχών, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο των έφιων μεταφορών στην Ευρώπη στο μέλλον, όπως υπόθηκε, κινδυνεύουμε να έχουμε όλο και λιγότερους πόρους. Άρα τους πόρους, τους λίγους που έχουμε στη μας θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε με πιο έξυπνο τρόπο. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε λεπτομέρειες ε, αργότερα. Θα διατυπώσουμε τις προτάσεις μας στο ΔΥΜ μέσω τροπολογιών. Αλλά προς το παρόν θα ήθελα να επανέλθω στο πρώτο σημείο εξωτερικές σχέσεις. Νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει και η ανάπτυξη των εσωτερικών μεταφορών, του συστήματος των εσωτερικών μεταφορών. Πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το σύστημα. Καλό είναι να μιλάμε για τις σχέσεις μας με τον έξω κόσμο των εισαγωγικών, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται εντός Ευρώπης, τι σχέσεις υπάρχουν και διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών το περίφημο αυτό tube transport. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις διάφορες δυνατότητες και να μην βασιζόμαστε μόνο στη συγκεκριμένη μορφή μεταφορών. Δεν θα πρέπει να έχουμε μια στενή ε, προσέγγιση, αλλά να λάβουμε υπόψη και άλλες ε, εξελίξεις που έχουμε στην ανάπτυξη αυτών των μεταφορικών συστημάτων. Αυτοματοποίηση. Είναι ένα σημείο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αναφέρθηκε άλλωστε. Αλλά διαπιστώνω ότι μας διαφεύγει ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το περπάτημα, το ποδήλατο. Είναι σημαντικό και αυτό, να κινούμαστε με τα πόδια με ένα ποδήλατο. Ίσως ήθιστε πιο πολύ στην Ολλανδία ή στη Φιλανδία να βλέπει κανείς ποδηλάτες ή πεζούς, αλλά πρέπει να μας απασχολήσει. Vielen Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πασέκολτ. Ολλανδός, λέω μιλητής. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον συνάδελφό μου για αυτή τη Λευκή Βίβλο. Ήδη είχαμε μία πρώτη συζήτηση ε, και τότε έτσι μίλησα πάρα πολύ γενικά. Δεν θα το ξανακάνω. Πάντως θέλω να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου κύριε Βαντεκάμ τα καταφέρατε πάρα πολύ καλά το να παραμείνετε στοχευμένος ε, στα θέματα που διακυβεύονται. Εμείς ε, όταν θα καταθέσουμε τροπολογίες, αυτό που λείπει, γι' αυτό θα το κάνουμε εξάλλου, είναι ότι δεν υπάρχει κάποια επίγουσα μορφή. Γιατί αν δείτε λιγάκι το μέλλον των μεταφορών, είναι ο μόνος μεταφορέας ε, ο οποίος ε, παρουσιάζει αύξηση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ε, όλοι είμαστε σε μια φάση να περιορίζουμε αυτές τις εκπομπές εκτός από τον τομέα των μεταφορών. Πρέπει λοιπόν να το θίξουμε αυτό το θέμα και πολύ πιο σκληρά. Και το δεύτερο, αυτή η μετατροπή του μοντέλου ε, που όλοι το λένε, αλλά αν δει κανείς λιγάκι την πραγματικότητα, αυτή η μετατροπή δεν λαμβάνει χώρα και άρα, εντάξει, μπορούμε να μιλάμε για όλα αυτά, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πιο αυστηρό ύφο και να διασφαλίζουμε ότι όταν ε, υπάρχει νέα αξιολόγηση του μέλλοντος των μεταφορών πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί από το να μιλάμε σε μια ανακοίνωση ότι οι μεταφορές είναι ένας ε, πολύ σημαντικός τομέας. Ε, δεν ισχύει αυτό στην περίπτωσή μας. Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε τροπολογίες και θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην αλλαγή του μοντέλου και τις ε, τιμολογήσεις ε, σε αυτά τα δύο θέματα. Γιατί αν δει κανείς λιγάκι το θέμα των τιμολογήσεων, κατά την άποψή μου θα πρέπει να είμαστε πιο προκλητικοί επί του θέματος ε, της τιμολόγησης. Γιατί εκεί είναι σαφές ότι παίζει ρόλο η τιμολόγηση, κυρίως στις οδικές μεταφορές. Και αν το κάνουμε με βάση τις, τα χιλιόμετρα, την χρήση των ε, δρόμων, να εστιάσουμε και στο θέμα του χρήστη, πρέπει να δούμε πώς ακριβώς όλα αυτά ε, τα οποία ε, χρησιμοποιούνται το κόστος της χρήσης των οδικών μεταφορών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επ' αυτού θα καταθέσουμε τροπολογίες. Και θα δούμε λιγάκι και τα διάφορα είδη μεταφορών. Νομίζω ότι και εκεί η γλώσσα μπορεί να είναι πιο αυστηρή. Γιατί αν δείτε λιγάκι το πώς ακριβώς τιμολογούμε τις, τα διάφορα είδη μεταφορών, ε, προκύπτει σαφής αδικία απόλυτη αδικία. Και ένας από, ένα από τα είδη μεταφορών είναι οι αερομεταφορές που εξαιρούνται από σχεδόν τα πάντα. Και αυτό λοιπόν πρέπει να το εξετάσουμε. Αν θέλουμε θεμητό ανταγωνισμό ανάμεσα στα διάφορα είδη μεταφορών, τότε θα πρέπει ε, τιμία να είναι και τιμολόγηση και να περιλαμβάνει ε, ξεκάθαρα το κόστος, την ε, αποκαλούμενη εσωτερικοποίηση του κόστους. Αυτό όμως δεν γίνεται και έτσι προκύπτει Αθέμητος ανταγωνισμός που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πιο σκληρά και γι' αυτό εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες. Και θα δούμε πιο συγκεκριμένα τις αερομεταφορές, διότι η φορολόγηση της κυροζήνης δεν αναφέρεται ή το ΦΠΑ στις αερομεταφορές, ούτε και αυτό. Όλες αυτές λοιπόν οι εξαιρέσεις δεν είναι σωστές και τώρα ε, ο ΙΚΑΟ ε, ξετάζει, αρχίζει ενδεχομένως ε, κάποια συμφωνία ίσως το 2020. Κοιτάξτε, δεν είναι σωστό αυτό. Έχει φτάσει η χρονική στιγμή να είμαστε πιο επιθετικοί. Εμείς λοιπόν θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό γιατί οι αερομεταφορές έχουν εξαιρεθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δεν είναι επειδή εγώ είμαι κατά των πτήσεων, αλλά όλοι να πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί και να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός. Και οι χρήστες των μεταφορών να έχουν μπροστά τους μία δίκαιη ε, επιλογή. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή οι αερομεταφορές ευνοούνται προκλητικά. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Βαντεκάμπ εξακολουθούμε να μην έχουμε καταλάβει πώς ακριβώς ε, θα οριστούν ε, δεσμευτικοί στόχοι μετά το 2020. Ο εισηγητής ε, προτείνει δεσμευτικό στόχο στις θαλάσσιες μεταφορές. Γιατί το κάνετε όμως αυτό μόνο σε αυτό τον τομέα. Με προβλημάτισε λιγάκι αυτή η πρόταση με την έννοια ότι εμείς θέλουμε δεσμευτικού στόχους στις μεταφορές αλλά γιατί μόνο στις θαλάσσιες μεταφορές. Αν θέλουμε να υπάρχει μια δίκαιη ίση κατανομή θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους. Με προβληματίζει λοιπόν γιατί προτείνεται αυτό το μέτρο μόνο για τις θαλάσσιες μεταφορές. Κατά τα άλλα, ε, στις ε, τροπολογίες ε, εμείς θεωρούμε ότι σε τελική ανάλυση υπάρχουν διεθνείς στόχοι για το κλίμα και για την βιοπικιλότητα και αυτοί πρέπει να τηρούνται. Γιατί μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι ε, ευνοούνται προκλητικά κάποια μέσα μεταφοράς και κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για την βιοπικιλότητα. Εμείς θα το δείξουμε στις ε, τροπολογίες μας γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν διεθνή πρότυπα και να σας υπενθυμίσω ότι στην ε, Διεθνή Συνθήκη για τη Βιοπικιλότητα λέμε ότι θέλουμε να διαφυλάξουμε τη βιοπικιλότητα. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν και εκεί κάποια μέτρα. Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα θέματα που θέλουμε να προσθέσουμε αλλά όπως σας είπα θα δώσουμε κυρίως σημασία στην εσωτερικοποίηση του κόστου ε, στην δίκαιη τιμολόγηση και στην αλλαγή του μοντέλου που πρέπει να λάβει η χώρα και όχι μετά από πέντε χρόνια όπου ο κύριος Βαντεκάμπ θα είναι εδώ για την ενδέκατη χρονιά του στο Κοινοβούλιο θα παρουσιάζει πάλι μια λευκή βίβλο για τις μεταφορές που θα λέει στο σωστό δρόμο είμαστε αλλά δεν έχουμε ακόμα πετύχει τους στόχους μας. Εμείς ελπίζουμε μετά από πέντε χρόνια να έχουμε να ε, παρουσιάσουμε από τα αποτελέσματα και ελπίζω ε, και ο κύριος Βαντενκάμπ ε, να προσβλέπει και αυτός στο να υποβάλει μετά από πέντε χρόνια μια τελείως διαφορετική έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Πίτερ Λούνκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόκειται για μια καλή, ισορροπημένη έκθεση. Αλλά μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα πράγματα. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ένα σωστό λειτουργικό σύστημα μεταφορών για την ενιαία αγορά. Άρα πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και το διοικητικό βάρος. Πρέπει να υπάρχει μια σαφής εικόνα όταν ε, υπάρχει κατάχρηση των κανόνων του καμποτάζ. Να δούμε την κατάσταση που υπάρχει ε, στο θέμα του ανταγωνισμού στις αερομεταφορές. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που έχουν ε, να κάνουν με τις εργατικές και κοινωνικές διαστάσεις, αλλά γενικά όταν επιβάζεις ε, κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκ των άνω προς τα κάτω υπάρχει πάντα ε, κίνδυνος καταχρήσεων. Οι καταχρήσεις, οι παρατυπίες του υφιστάμενου συστήματος προστατεύονται από τους κανόνες αυτή τη στιγμή. Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Τώρα, για το, το κοινωνικό dumping που δημιουργείται από το, το κυνήγι του κέρδους. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία οι ανεμβίαστοι χειριστές είναι αυτοί που αλλάζουν ε, τους κανόνες προς όφελός τους πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πολύ πιο αυστηρή νομοθεσία που θα αντιμετωπίζει σωστά όλους εκείνους τους επιχειρηματίες του χώρου που λειτουργούν χωρίς ε, ενδιασμούς. Και νομίζω ότι το κείμενο αυτό θα αποτελέσει μια ευκαιρία όλοι να μπορέσουμε να ε, ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μειώνοντας τις καταχρήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές ήταν ε, οι παρεμβάσεις του εισηγητή και των σχεδόν εισηγητών. Έχουν ζήσει το λόγο πάρα πολύ και πρέπει να περιοριστείτε σε δύο λεπτά. Το λόγο έχει κύριου κύριος Νίλσεν για δύο λεπτά. Ε, θα είμαι σύντομος. Πολύ καλή έκθεση, ισορροπημένη σημαντικό να δώσουμε ότι οι βιώσιμες μεταφορές έχουν να κάνουν και με την εργασιακή βιωσιμότητα, όχι μόνο με την οικολογική. Μην ξεχνάτε ότι το Σεπτέμβριο ψηφίσαμε ένα ψήφισμα με πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που θεωρούσε ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ έπρεπε να καταργηθεί. Διότι φεύγουν από την αγορά οι σοβαρές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή είπε τώρα ότι ε, θέλει να αναθεωρήσει τους κανόνες για το καμποτάζ. Πρόκειται για μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Η έλεγχοι πρέπει να γίνονται από το κράτη-μέλη. Όταν ε, μιλούμε για τις αερομεταφορές έχουμε χρόνο να δούμε πώς τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν μεταξύ καινοτόμων επιχειρήσεων, ε, εταιριών κατασκευής και χωρίς να υπάρχει μείωση της ασφάλειας πτήσεων. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε ταυτόχρονα. Η ασφάλεια πρέπει να είναι σαφέστερη στην έκθεσή μας. Επίσης πρέπει να δούμε τους βασικούς κανόνες του ICAO. Εάν γίνει κάτι τέτοιο θα βελτιωθεί και η ασφάλεια γιατί πιστεύω ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των συνθήκων απασχόλησης και πρόσληψης και της ασφάλειας. Πολυτροπικότητα, περιβάλλον, δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικό επίσης. Κάτι άλλο. Είμαι εκπρόσωπος για τον τομέα των μεταφορών και της προσλήψης. Και εδώ πρέπει να ε, δούμε την κατάσταση προσεκτικότερα. Στον τομέα των μεταφορών δουλεύουν πολλοί άντρες, πολύ λιγότερες γυναίκες. Ευχαριστούμε πολύ. Κριστίν Ρεβονταλό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να σεβαστώ το χρόνο που μου δώσετε. Πολλά από αυτά που περιέχει η έκθεση είναι σωστά. Ο στόχος του εισηγητή είναι να έχει μία προσέγγιση για την ενίσχυση των μέσων και τον καθορισμό νέων στόχων είναι μια καλή ευκαιρία για την επιρροή στην ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η διατροπική μετα, μετακίνηση και η εφαρμογή της αρχής, ο, ο και ο χρήστης πληρώνουν, είναι λογικό και ότι πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα και στην τιμολόγηση και στις υποδομές. Χωρίς η ισχυρή πολιτική δέσμη στον τομέα αυτό, η Ένωση δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της. Στη φάση αυτή καμία νομοθετική πρωτοβουλία δεν πρέπει να αποκλειστεί μέχρι το 2030 πρόκειται για έναν φιλόδοξο στόχο που θα πρέπει να λειτουργήσει προ όφελο των δημοσίων ε, μεταφορών. Επίσης, εκφράζω την ικανοποίησή μου για τις προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπομπή ε, διοξιδίου του ανθρώπου από τα βαρέα οχήματα. Ωστόσο, πολλά θέματα πρέπει να τεθούν. Πρώτον, αναφέρθηκε από τον συνάδελφο Γέννη το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το ρόλο των μεταφορών ως παράγοντα κοινωνικής ένταξης, η προσβασιμότητα των μεταφορών, το δικαίωμα στην κινητικότητα, η προτεραιότητα των δημοσίων ε, μεταφορών ως τρόπος καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να είναι στοιχείο της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής μας. Η αναγνώριση της υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσία για να εξασφαλίσει μια ε, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις καλύτερε προποθέσει είναι μια θεμελιώδης ε, δέσμευση που δεν πρέπει να χαθεί στη Λευκή Βίβλο. Τέλος, η δημιουργία ενός κοινωνικού κώδικα για την ε, κινητικότητα πρέπει να συζητηθεί, είναι ενδιαφέρουσα ιδέα και πρέπει να συζητηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους με σεβασμό ωστόσο των εφιστάμενων ευρωπαϊκών κανόνων. Εντάχει, πρέπει να μεταφερθούν σε νομοθετικά κείμενα οι στόχοι του, της Βίβλου για τη μείωση κατά 60% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Πολύ ωραία. Από κοινού ε, χρησιμοποιήστε τέσσερα λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, ο κύριος Μπαχ, λέει κύριος Μπαχ, και εγώ ευχαριστώ πολύ τους συγητές και επίσης ε, θέλω να πω ότι και εγώ το συγχαίρω, όπως και οι προλαλήσαντες ε, Ετήγησαν ε, διάφορα θέματα, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, γι' αυτό θα εστιάσω την προσοχή μου σε τρία-τέσσερα θέματα. Καταρχήν όσον αφορά την πολυτροπικότητα που αυτό θα γίνει όλο και πιο σημαντικό, ε, θα είναι η συνλειτουργία ε, των ε, διαφόρων μέσων μεταφοράς. Αυτά που είπε και ο συνάδελφος Κοκ για το ticketing και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, να ζητήσουμε από την Κομισιόν να λάβει υπόψη της την κατάσταση που υπάρχει σε όλα τα μέσα μεταφορών και την εναρμόνιση των ε, νομικών και νομοθετικών διατάξεων. Στα κράτη-μέλη να γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων, να, αναλυθεί, να αναλυθούν οι επιπτώσεις και με βάση την αναλύση, ανάλυση που θα προκύψει να κατατεθεί και μία πρόταση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει διολίστηση προς τα κάτω, στο σύνολο των μεταφορών. Στις αερομεταφορές, στις, στους σιδηρόδρομους, στις οδικές μεταφορές έτσι και αλλιώ. Ε, εκτός από τις ε, κοινωνικές συνθήκες υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας. Κατόπιν, ε, τα δικαιώματα των επιβατών. Και στο θέμα αυτό έχω κάθε κατανόηση Υπάρχουν ε, μεμονωμένες εκθέσεις και προτάσεις της Επιτροπής ε, για τα διάφορα είδη μεταφορών. Σε γενικές γραμμές πάντως ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Να υπάρχει ένα έδος χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των επιβατών όσον αφορά την αποζημίωσή τους, την ενημέρωσή τους. Να υπάρχει λοιπόν ένα σφαιρικό πλαίσιο για να υπάρχει και δικαιοσύνη ανάμεσα στα διάφορα είδη μεταφορών. Τώρα, ε, για τις αερομεταφοτερές ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, κυρίως και για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία στο άμεσο μέλλον θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα των υποδομών. Σας ευχαριστώ πολύ. Dziękuję Ευχαριστώ πολύ κύριε Θέλω καταφέρω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω Θέλω καταρχά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλο και Παράτσκη τον εισηγητή για την πολύ καλή του δουλειά. Κάποιε παρατηρήσεις, αν με επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα, στο σημείο C, λέτε ότι είμαστε παγκόσμιοι για στον τομέα των μεταφορών. Ακόμη. Θα έπρεπε να λέει. Εξακολουθούμε να είμαστε δηλαδή ηγέτες. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο τομέας μεταφορών για την ε, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Τι θέλω να πω. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. Οι μεταφορές σίγουρα υποτίθεται ότι πρέπει να πρέπει να βελτιώνουν και το βιωτικό επίπεδο. Άρα εκεί θέλουμε πιο πολλά στοιχεία. Το πλήρω ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, στο D. Έχω το εξή ερώτημα. Η γαλλική και ε, γερμανική φόρη. Αυτά τα τέλη, 8 με 9 ευρώ για τι μεταφορέ. Τι κάνουν, βελτιώνουν την κατάσταση ή όχι. Έχουμε ένα έγγραφο το οποίο καλά τα λέει, αλλά από την άλλη έχουμε και την πραγματικότητα. Αυτά που γίνονται στην πράξη. Τι κάνουν οι κυβερνήσει, ε, το κράτο για την πολιτική μεταφόρων και συγκοινωνιών. Πρέπει να σχολιάσουμε και αυτά. Σίγουρα η Λευκή Βίβλος ε, είναι δεσμευτική για τα κρατημέλη ή μήπω δεν είναι, άρα ολοκληρωμένε μεταφορέ. Εδώ τι έχουμε. σε πρόσβαση στι συνδρομικέ μεταφορέ κτλ. Αυτά όμω που προβλέπονται παρακολύουν την καλή τον καλό συνδυασμό συνδρομικών μεταφορών με άλλους τρόπους μεταφοράς. Το σχέδιο Juncker τώρα είναι πολύ καλό στο 7 αυτό που λέγεται ως δυνατότητα όμως possibility. Αλλά στο 7 πώς θα γίνει δυνατό αυτό. Τι θα κάνουν τα κράτη, θα κάνουν κυβερνήσει, γιατί και από αυτέ εξαρτώνται πολλά. Πάντω το έγγραφο είναι καλό. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, να τον συγχαρώ και με τι τροπολογίε μα ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πράξει τα δέοντα. Γιατί μεταφορέ είναι προτεραιότητα ω ευρωπαϊκή πολιτική και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσει και η Κομισιόν. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Κοχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Βίμ, σε συγχαίρω για την πολύ καλή σου εισήγηση. Τρει παρατηρήσει θα κάνω. Ε, πολύ καλά τον τομέα των μεταφορών ω ε, οικονομικό τομέα, αλλά για μένα ρόλο παίζουν τα δικαιώματα των επιβατών, κυρίω των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. Να βοηθήσουμε την ασφάλεια να υπάρχει υπάρχουν δομές που να μπορούν να τις πληρώσουν οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν αναπηρία. Υπάρχει και το θέμα των υποδομών. Ε, βεβαίως και είναι σημαντικό ε, να υπάρχει βιώσιμος σχεδιασμός, ε, ευθύης διασύνδεση των μεταφορών με τις μονάδες και τις διαδικασίες παραγωγής. Το τρίτο που παίζει ρόλο είναι το όραμά μας για το αυτόνομο ή το ημι αυτόνομο οδήγημα, την αυτόνομη αυτό δεν είναι πολύ σαφέ, ίσω πρέπει να το κουβεντιάσουμε λιγάκι αυτό. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρο, επόμενο ομιλητή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ο κύριο Ερτούκ, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή. Ε, πολύ καλή η έκθεσή του, διότι στην έκθεσή του θίγει πολλά και σημαντικά θέματα. Θα ήθελα να αναφέρω τα εξή ε, σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα των δύο λεπτών που έχω στη διάθεσή μου. Βρίσκω πολύ καλό και σημαντικό να ε, αναφέρονται τιμές ε, που προβλέπονται για το μέλλον. Επίσης η προαγωγή ε, της βιώσιμης κινητικότητας και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι η ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων, TNT. Αυτό που διάβασα με εξέπληξε ήταν ο στόχος για το διπλασιασμό των χρηστών των δημόσιων μέσων μεταφοράς ε, μέχρι το 2030. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, πράγματι πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες, καλώντας τα να επενδύσουν στις δημόσιες μεταφορές. Γιατί αν θέλουμε το διπλασιασμό του αριθμού των χρηστών, που το θέλουμε όλοι μας, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς ε, περαιτέρω επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων μας και αυτό επίσης ε, που με χαροποίησε πάρα πολύ ήταν ο κοινωνικός ε, κώδικας ε, για τους επαγγελματίες οδηγούς το 2016. Αυτό θα αναφέρεται στο Road Package. Είναι λοιπόν σημαντικό. Και υπάρχει και κάτι άλλο καθοριστικής σημασίας, δηλαδή ανάμεσα στην πολυτροπικότητα την οποία υποστηρίζω ανεπιφύλακτα γιατί η πολυτροπικότητα σημαίνει βελτιστοποίηση ενός ε, είδους μεταφοράς με την χρήση και άλλων. Κατά την άποψή μου όμως ε, αυτός δεν είναι ο κυρίαρχος στόχος ε, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει άλλους δεσμευτικούς στόχους, δηλαδή τα εμπορεύματα να μεταφερθούν στους σιδηρόδρομους, ο κανόνας των 300 χιλιόμετρων. Επ' αυτού θέλω να μας διευκρινίσετε ε, τι ακριβώς έγινε και με όλα τα άλλα που προτείναμε στη Λευκή Βίβλιο του 2011. Η Όλγα Σελένοβα, επόμενη μιλήτρια. Παρακαλώ. Ε, Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω για τη Λευκή Βίβλο του 2011. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνεται να αναλύσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους που ανέφεραν ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι εργασίες, οι συνθήκες εργασίας όσων εργάζονται στον τομέα των μεταφορών. Και τώρα τρεις συγκεκριμένε παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Υποθέτω ότι έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό καθήκον και αυτό αφορά στις ε, αποστάσεις, διαφορετικές αποστάσεις ε, στα κράτη-μέλη. Βεβαίως αυτό έχει σχέση με την ε, εδαφική συνοχή και οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Και το θέμα της ασφάλειας. Πράγματι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια με τη λήψη πολλών μέτρων και με τη νέα τεχνολογία. Όμως αν επιτιμούμε οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν περισσότερο τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς, κυρίως στις πόλεις, τότε πρέπει να διασφαλίσουμε οι μεταφορές να είναι βιώσιμες όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στις ε, υπεραστικές μεταφορές. Να υπάρχουν και ασφαλείς δομές και για ε, ποδηλάτες και για τους πεζούς και κάτι που ξεχάστηκε. Δηλαδή η έκθεση δεν ενδιαφέρει, δεν αναφέρει τα ανοιχτά λεωφορεία τα οποία υπάρχουν στις πόλεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κλούν. Να ευχαριστήσω το ΒΙΜ, γιατί έχουμε χάρη στη δουλειά του μια πολύ ξεκάθαρη έκθεση αναχείρας. Και όπως είπε και ο ίδιος, ουσιαστικά πρόκειται για μια αξιολόγηση του, της Λευκής Βίβλου. Καιρός είναι να δούμε λοιπόν τι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και πού μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις με στόχο να εκμεταλλευτούμε τις τεχνολογικές προόδους, την καινοτομία, αστικές μεταφορές, Άλλωστε, σε αστικά κέντρα ζει το 80% του πληθυσμού, άρα είναι σημαντικέ οι αστικέ μεταφορέ. Και οι οδικέ μεταφορέ και το περπάτημα, βέβαια, και το ποδήλατο, οι δημόσιε συγκοινωνίε και αυτά είναι θέματα σημαντικά και τα καλύπτει πολύ καλά ο Βίμ στην έκθεση στον τομέα ε, των αερομεταφορών. Νομίζω ότι εκεί μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Υπάρχουν ε, στοχίες και αποτυχίες ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Εδώ πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ανταγωνιστικότητα. Δεν έχει υπάρξει σωστή εφαρμογή, πραγματικά περί αποτυχίας πρόκειται και αν δούμε τον ανταγωνισμό από τα κράτη του κόλπου θεωρώ ότι είναι σημαντικό η αναφορά αυτή που έγινε στον διάλογο για τα θέματα της αεροπορίας. Τώρα, δίκαιος ανταγωνισμός. Ετέθηκε αυτό το θέμα, το συζητήσαμε. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, και το είπαν άλλοι προλαλήσαντες, ότι δεν είμαστε αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν πτυχές, κοινωνικές, ε, εργασιακά ζητήματα, κρατικές ενισχύσεις, ε, στήριξη αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρεών από κυβερνήσεις που δεν ελέγχονται ούτε από την Κομισιόν ούτε από τα κράτη-μέλη, μάλλον από εμάς. Άρα ο διάλογος αυτός θα είναι σημαντικός. για το βιβλίο η οι άλλες ευρωπαϊκές εταιρείε του κόλπου, τα ερωμένα μοιράτε κτλ. έχουν πολύ έντονη παρουσία ε, στο Δουμπλίνο. Μεταφέρουν επιβάτες ε, προς Ανατολάς, ε, προς την Ανατολική Ασία. Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν με πολύ μεγάλη χαρά τις εταιρείε αυτές. Είναι πρόκληση, αλλά με το διάλογο νομίζω μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο και γενικά και στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών έχουμε αυτή τη δυνατότητα των θαλάσσιων αυτοκινητοδρόμων. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε γιατί δεν έχουμε ακόμη εξοπλίσει επαρκώ αυτέ τι δυνατότητε, ιδίω σε διασύνδεση οδικού δικτύου με λιμένε μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων. Ευχαριστώ. Ντέλη. Ευχαριστώ. Την ε, τελευταία φορά όταν είχαμε ανταλλαγή απόψεων επισήμανα ότι την έκθεση αυτή την ε, θεωρώ ισόρροπη. Και δεν θέλω να σπαταλήσουμε το χρόνο μας, ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο θέματα. Το ένα είναι, μου αρέσει πάρα πολύ, το ότι η έκθεση αυτή προβάλλει τον ανθρώπινο παράγοντα Κατόπιν τούτου είναι σημαντικό να προβάλλουμε ότι έχουν μεγάλη σημασία οι εργασίες της Κομισιόν, δηλαδή το νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και ίσως στην έκθεση θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτοί οι κανόνες ε, πρέπει να είναι διαφανής και επίσης ε, είναι σημαντικό οι κανόνες να παραμείνουν και προβλέψιμοι. Αυτό μπορεί να βοηθήσει και την καινοτομία και τις επιχειρήσεις. Τώρα το σύστημα της ε, πιστοποίησης είναι πολύ σημαντικό και εξίσου σημαντικό είναι τα πάντα να παραμείνουν προβλέψιμα. Αυτό... Τι λοιπόν, αυτό είναι ένα αίτημα προς την Επιτροπή. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά στην ε, ε, διεύρυνση των υποδομών. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την έκθεση και απλά ε, θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα σημειολογικό. Στα αγγλικά υπάρχει όρος missing link, αλλά εδώ θα πρέπει να μιλάμε για bottleneck, για ε, στενοπό αν θέλετε. Αυτή τη λέξη, αυτόν τον όρο στενοπό, το bottleneck, δεν τον βλέπω να υπάρχει στην έκθεση. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το τι γίνεται στη γειτονιά μας. Τα αντιευρωπαϊκά δίκτυα είναι σημαντικά και για τις γειτονικέ χώρες πρέπει αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Επόμενος ομιλητής, Μάτις Φον Μίλτενμπεργκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να συγχανώ και τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά τους. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Στην έκθεση αυτή το σχέδιο έκθεσης είναι, γίνεται έκκληση να υπάρξει διάλογος με τις χώρες του κόλπου, να υπάρχουν διαφάνειες τις ενισχύσεις, να υπάρχει θεμητός ελογονισμός. Κύριε Ισηγητά, γιατί δεν μιλάτε για την Τουρκία, όχι μόνο λόγω της σημασίας της χώρας, ε, είναι μια αγορά μεγάλη, γειτονική, αυξάνεται, σημαντική για μας. Τι γίνεται εκεί με την ανάπτυξη των, υποδομών του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης. Εκεί πρέπει να υπάρχει οικονομική διαφάνεια και θεμητός ανταγωνισμός. Γιατί λοιπόν δεν αναφέρεται η Τουρκία στην έκθεσή σας. Ελπίζω η Κομισιόν πιο μετά να παρουσιάσει νέες προτάσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων των αερομεταφορών στην Ευρώπη. Να μην λειτουργούμε μόνο αμυντικά έναντι των χωρών του κόλπου, αλλά να υιοθετήσουμε μια πιο ε, διενεργή στρατηγική, πιο αισιόδοξη στρατηγική για να κερδίσουμε νέες αγορές στην Ασία. Η αύξηση των ε, ε ταξιδιωτών γίνεται, των επιβατών γίνεται κυρίως στην Ασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιζελιέ, εκτός μικροφώνου. Ναι, εκτός μικροφώνου μιλητής. Και εγώ όπως και όλοι οι συνάδελφοι να συγχαρούμε τον εισηγητή για την δουλειά που έκανε. Επιτυχώς και με συνθετικό τρόπο. Δεν θα προσθέσω πολλά. Απλά να εκφράσω μια, ε, ένα παράπονο. Γίνεται λόγος στον έντονο ανταγωνισμό, αλλά όχι επαρκώς. Το, η Λευκή Βίβλος το είχε, η έκθεση το αναφέρει αλλά δεν το υπογραμμίζει. Μιλώ λοιπόν την ανάγκη να υπάρξει ανταγωνισμός βάσει σαφών αρχών. Προφανώς είναι σημαντική η αμοιβαιότητα στον τομέα αυτό. Να μετέχουν όλοι στις δικές μας αγορές εφόσον οι δικές μας επιχειρήσεις μετέχουν στις αγορές των άλλων. Ένα θετικό επίσης που είναι πιο λιγότερο πολιτικό. Εμείς μιλάμε για το 2050 σαν χρονικό ορίζοντα μιλώντας για τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτό. Ωραίο. Εγώ δουλεύω όμως με τα drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μην ξεχάσουμε λοιπόν μια τεράστια εξέλιξη που γίνεται σε ό,τι αφορά την αυτοματοποίηση των μεταφορών. Οχήματα που περνούν από την ανθρώπινη στην αυτόματη οδήγηση. Το Ρότερνταμ που γνωρίζει ο εισηγητής καλά έχει ξεκινήσει να μελετά το θέμα της αυτοματοποίησης. Πρόκειται για ένα σημαντικό τομέα στο μέλλον πρέπει να υπάρξει μια μελέτη για τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης των μεταφορών που έχει πολλές επιπτώσεις. Πολύ ωραία. Εγώ είμαι ο τελευταίο ε, που είχα ζήσει λόγο. Ε, προφανώς Προφανώ και ευχαριστώ τον κύριο Βαντενκάπ για την εισήγησή του. Ε, Στη συζήτηση όμως ε, θέλω να υπογραμμίσω το εξής, ότι όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς ε, υπάρχει άδικη μεταχείριση. Ευνοούνται αυτοί που βλάπτουν το περιβάλλον και τα μέσα τα φιλικά προς το περιβάλλον επιβαρύνονται υπέρμετρα. Αντικία υπάρχει και όσον αφορά στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάναμε κάποια ανάλυση στα διατροτικά ταμεία 60% στον δρόμο, ε, το 30% στο, στους πρόδρομους και τα υπόλοιπα μόνο σε άλλα μέσα. Έτσι όμω δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πετύχουμε τους στόχους μας του κλίματος γιατί αν επενδύουμε σε λάθο κατεύθυνση ε, δεν θα έχουμε αρκετά χρήματα. Άρα δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταθέσει ένα σχέδιο το πώς θα τα περιορίσει όλα αυτά. Βεβαίω και γνωρίζουμε ότι η επικορικότητα είναι πολύ σημαντική αλλά πρέπει να ακολουθείται σωστό δρόμο. Στο Ελσίνκι υπάρχουν μελέτες ε, όπου ένα ευρώ στα ποδήλατα φαίνουν πίσω 8 ευρώ αν λάβει κανείς υπόψη του τα νοσοκομεία και όλα τα άλλα. Οικονομικά λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η λύση και όχι μόνο οικολογικά και αυτή θα πρέπει να είναι η σωστή κατεύθυνση. Το 70% των εκπομπών που βλάπτουν το περιβάλλον έρχονται από αυτά τα μέσα μεταφοράς και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω τους δισταγμούς που υπάρχουν σε σχέση με το model shift. Υπάρχουν φανταστικά παραδείγματα. Είχαμε την ακρόαση για την κινητικότητα Αναφέρθηκε λοιπόν ότι υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα τα οποία απλά χρειάζεται να μιμηθούμε. Ένα θα αναφέρω, Κοπενχάγη σε 20 χρόνια θα υπάρχει αύξηση κατά 300% στα, στα Σήμερα ένας τεράστιος αριθμός ε, ανθρώπων στην Κοπενχάγη πάνε στη δουλειά τους στα πανεπιστήμια με το ποντήλατο. Αν τους το είχαν πει πριν από 20 χρόνια θα έλεγαν ε, καλά ε, τι λέτε, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Αλλά να, υπάρχει θετικό παράδειγμα. Ακόμα και στο Βερολίνο ε, υπάρχει μεγάλη αύξηση στα ποντήλατα. Ακόμα και στη Σεμπίλια έχουμε πολύ καλά παραδείγματα παραδείγματα στη Νότιο Ισπανία. Άρα δηλαδή όλα αυτά μπορούν να γίνουν, έχουμε καλά παραδείγματα και χρειάζεται απλά να τα μιμηθούμε. Αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση και δεν καταλαβαίνω γιατί διστάζεται στο model shift. Σημαντική η πολυτροπικότητα, αλλά το model shift είναι πιο σημαντικό να περάσουμε ε, στο ποδήλατο και στην ε, πεζοπορία γιατί ε, πολλές αποστάσεις στις πόλεις είναι μικρότερες από 6 χιλιόμετρα. Αυτές είναι καλές αποστάσεις για το model shift. Πολύ ωραία και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Ολιβιέ Ονίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε. Καταρχά να σα ευχαριστήσω για τι ψηφοφορίε σήμερα το πρωί για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Πρόκειται για μια σημαντική συμβολή από πλευρά σας που ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στη διαδικασία συναπόφασης ώστε να είναι απόλυτα συμπληρωματικό το ταμείο αυτό με τα άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ως το μέτρο του δυνατό. Για τη Λευκή Βίβλο, εγώ δεν θα έλεγα ότι η έκθεση του κυρίου Βαντερκάμπ είναι κάπως, και κάπως έτσι, κάπως αλλιώς. Μια εμπειρία του κυρίου Βαντερκάμπ είναι ακριβώς η ποιότητα της ε, συμβολής του και που εκφράζει και την ποιότητα της συμβολής της Επιτροπής. Σήμερα το πρωί είδαμε ότι η έκθεση κερδίζει και θα αποκομίσει περισσότερα προς βελτίωσή της από τις ιδέες των μελών της Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι έχει μια στεναρή, σωστή ανάλυση και πολύ σοφή προσέγγιση. Η έκθεση δεν ε, επιχειρεί να αλλάξει το σύστημα, αλλά να δώσει έμφαση στην συνέχεια και την εφαρμογή αυτών που πρέπει να εφαρμοστούν με συγκεκριμένες εμφάσεις. Περιλαμβάνει νέες διαστάσεις που είτε διορθώνουν πράγματα που υποτιμήθηκαν στο παρελθόν. Φέτος, για παράδειγμα, ε, εμφανίζεται εντονότερη κοινωνική διάσταση ή που έχουν στόχο να προσαρμόσουν και να ενημερώσουν τις πρωτοβουλίες της Λευκής Βίβλου, στις ταχύτατες εξελίξεις, ιδίως στον τομέα των νέων υπηρεσιών και των τεχνολογικών εξελίξεων. Από πλευράς μας θεωρούμε ενδιαφέρον να υπάρξουν περαιτέρω μηνύματα και ιδέες σε κάποιους τομείς. Για παράδειγμα, κάποιοι τονίσατε την εξωτερική διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Κάτι πολύ σημαντικό. αλλά όχι μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά και σε τι βαθμό έχουμε δίκαιη πρόσβαση σε άλλες αγορές, παρέχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση στην δική μας αγορά προς τρίτες χώρες μάλλον προς επιχειρηματίες τρίτων χωρών. Επίσης, έμφαση στην ολοκλήρωση κάποιων συνεχιζόμενων φακέλων, π.χ. ο σιδηροδρομικός τομέας. Εδώ κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά για να ολοκληρωθεί το τέταρτο πακέτο σιδηροδρομικών μεταφορών. Πιο σημαντικό δε να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο των λιμένων που θα είναι κρίσιμη, που είναι και θα είναι κρίσιμη παράγοντες στη σημερινή οικονομία και καλύτερη σύμμαχοί μας για την ολοκλήρωση της αλυσίδας επιμελητίας στην Ευρώπη συνολικά. Άλλη διάσταση, κοινωνική. Δεν περιμένουμε βέβαια οι μεταφορές να δημιουργήσουν εργατικό δίκαιο, αλλά αν η έκθεση μας βοηθήσει να ενισχύσουμε κάποιες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση των συνθήκων εργασίας των, ε, του κλάδου των μεταφορών και την ελκυστικότητα του τομέα αυτού για τους εργαζομένους θα ήταν κάτι εξαιρετικά θετικό. Το ίδιο και θα βοηθούσε να εξασφαλίσουμε δίκαιες συνθήκες μεταξύ των κλάδων. Αεροπορικά πρώτα-πρώτα, τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών που θα αναθεωρηθούν σημαντικά φέτος και των οδικών που όπως σημειώσατε θα περάσουν θα ενταχθούν σε ένα μεγάλο πακέτο νομοθετικών προτάσεων του χρόνου. Ε, η άλλη διάσταση της βιωσιμότητας που εκτιμήσαμε στην έκθεση ιδιαίτερα είναι το ότι κοιτάζει την έννοια της βιωσιμότητας ε, από γενική, ε, από μια σφαιρική προσέγγιση και τις υποδομές και τη συντήρηση και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο πρωτοβουλειών για τη βελτίωση της ασφάλειας τόσο ενεργητικής όσο και παθητικής, παράγοντες που επηρεάζουν την ε, βιωσιμότητα, η αποτελεσματικότητα της ενέργειας, και εδώ είναι κάτι σημαντικό, κάποιοι τομείς όπου χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα και βεβαίω την διάσταση των αστικών μεταφορών. Πολύ το τονίσατε σήμερα. Μια άλλη τέταρτη διάσταση. Καινοτομία. Τα έξυπνα συστήματα, όπως τα περιγράφει το κείμενο. Εδώ πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην προσέγγιση της, της συνολικής ε, κινητικότητας από πόρτα σε πόρτα, ενισχύοντας την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Πολλά ζητήματα έχουν να κάνουν με τη διαλειτουργικότητα, μόνιμη προτεραιότητα της Ένωσης στον τομέα των ε, μεταφορών και μια πιο μεγάλη έμφαση στην, στις αυτόματες μεταφορές, αν θέλουμε να έχουμε μια, να διατηρήσουμε την παγκόσμια ηγεσία μας στον τομέα των μεταφορών, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην αυτοματοποίηση. Το κάναμε στις αερομεταφορές με το ΣΕΖΑΡ. Στους άλλους κλάδους ωστόσο έχουμε μια πιο δειλή προσέγγιση. Θα ήταν καλό να υπάρχει λοιπόν μια ισχυρότερη προσέγγιση στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα το λόγο έχει και πάλι ο εισηγητής. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίω είναι πάρα πολύ ευχάριστο το να εισπράττει κανείς ε, τόσες πολλές ε, φιλοφρονήσεις. Αλλά οι φιλοφρονήσεις ε, υποχρεώνουν αυτόν που τις δέχεται να ακολουθήσει σαφέστερη γραμμή Δυστυχώς ο συνάδελφός μου από το ECR, από το κόμμα αυτό, έφυγε, αλλά να επενθυμίσω ότι ζήτησε να υπάρξει μετατρέψη αντιμετώπιση ή μάλλον ελάφρυνση των στόχων βιωσιμότητας ε, και μετά έρχεται ε, εκπρόσωπος των Πρεσίων και λέει όχι μόνο δεν είναι σωστό αυτό αλλά οι ε, στόχοι της βιωσιμότητας πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί. Η δική μου λοιπόν η έκθεση προσπαθεί να βρει συμβιβασμό ανάμεσα σε όλα αυτά. Όλες οι πλευρές επιθυμούν να αποκτήσουν κάτι και ε, όσον αφορά τις τροπολογίες παρακαλώ ε, να μην ε, καταθέσετε 300 τροπολογίες αλλά 50 και αυτές να είναι στοχευμένες που νομίζω μπορεί κανείς να τις περιλάβει πολύ εύκολα στην έκθεση. Η Κλάντιο Ταπαρντέλα έχει απόλυτα δίκιο Πράγματι, κάπως ε, στην εισαγωγή μου δεν αναφέρω ιδιαίτερα τις αναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ε, Παραδείγματο χάρη την χρήση των υδάτων. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες ε, καινοτομία και θα το προβάλλω στην έκθεση. Ε, τώρα, πεζοί και ποδηλάτες. Οι ποδηλάτες πρέπει να στηριχθούν και οι πεζοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην Ολλανδία θεωρούμε ότι ε, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα στον τομέα αυτό και παράλληλα να ε, προστατεύεται και η ιδιωτική σφαίρα. Και η να Μάισνα έθεσε το θέμα πώς ε, μπορούμε να προστατεύσουμε την ε, ιδιωτική σφαίρα. Ε, και θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν χρησιμοποιεί κανείς δημόσια μέσα μεταφοράς, αυτό είναι λιγάκι δύσκολο, διότι όταν χρησιμοποιούνται τα δημόσια μέσα μεταφοράς ο χρήστης χάνει λιγάκι την ιδιωτική του σφαίρα και το έχουμε συζητήσει αυτό. Υπήρξε μία συζήτηση σχετικά με την επιβολή προστήμων διασυνοριακά. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι σημαντικά. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μία ένωση ε, και αυτό νομίζω ότι τη, διευκολύνει την ε, ε, προστασία των ε, δεδομένων. Κάτι άλλο που είπε επίση η Γκεζίνε για τις αερομεταφορές πράγματι, αυτό που είπε θα πρέπει να το λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας. Εκεί όμως όπου δεν έχω σκεφτεί ακόμα το τι θα κάνουμε είναι σχετικά με τις στοχευμένες επενδύσεις. Παραδείγματο χάρη μπορεί κανείς να μιλήσει για τα ασφαλιστικά ε, συμβόλαια. Αυτά να αντιοχετεύονται στις μεταφορές ή τα διόδια, ε, της εισπράξης από τα διόδια. Πάντως καταλαβαίνω τι θέλει να πει η Κιζίνε. Κοιτάξτε, εγώ έχω ένα αυτοκίνητο και για μένα αυτό παραμένει ένα μέσο χειραφέτησης. Ε, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν λιγότερα αυτοκίνητα στην πόλη, αλλά τι συμβαίνει με την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και ας δούμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Τουρκία. Ε, βλέπει κανείς ε, από πρώτο χέρι τι προβλήματα προκύπτουν με τόσα πολλά αυτοκίνητα. Αλλά τι γίνεται με τους ανθρώπους στην Ήπεθρο. Εκεί δεν είναι δυνατόν να τιμωρήσουμε τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Αυτό θα ήταν ανόητο. Κατόπιν ετέθη το ερώτημα γιατί μόνο οι θαλάσσιες μεταφορές. Κοιτάξτε, πρόκειται για στόχους ε, βιωσιμότητας και οι αερομεταφορές είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν ε, διεθνείς ε, συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή. Θεωρώ ότι δεν ζούμε σε ονειρεμένο κόσμο. Η Ευρώπη κατά κάποιον τρόπο ιστερεί Νομίζω ότι το έχουμε πει αυτό, χρειαζόμαστε ακόμα πιο καθαρούς ε, κινητήρες ε, που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, κατόπιν, σχετικά με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι συνάδελφοι που έθεσαν το ερώτημα έφυγαν. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Οι αστικές μεταφορές είναι τομέας υπευθυνότητας των κρατών μελών σε πάρα πολλές χώρες ε, διαπιστώνουμε ότι όταν τα πράγματα πάνε καλά ε, τα κράτη επέρονται και όταν κάτι δεν πάει καλά ε, αυτό μετακυλίουν το βάρος στις Βρυξέλλες. Άρα πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στις αστικές μεταφορές. Αυτό είναι θέμα επικουρικότητας και σαφώς και μπορούν να δραστηριοποιηθούν τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά αυτά τα λεωφορεία Αυτά τα λεωφορεία με ενδιαφέρουν ε, πάρα πολύ, αλλά ε, το θέμα της ιστορίας με την Τουρκία που ανέφερε ο συνάδελφος, ε, σωστά το είπε, ασχοληθήκαμε με την Emirates και την Etihad. Μας φιλοξένησε Turkish Airlines που μας παρουσίασε όλα τα πλεονεκτήματά της. Αυτό όμως που ελέγχθη σε σχέση με την Τουρκία είναι σωστό. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για τις ε, παρατηρήσεις της ε, και περιμένουμε τώρα τις ε, τροπολογίες. Παρακαλώ όμως να μην καταθέσετε τόσο πολλές τροπολογίες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον εισηγητή και όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Έτσι λοιπόν για σήμερα το πρωί κλείνει η δημόσια συνεδρίαση και περνάμε στη συνεδρίασή μας και κλεισμένων των τυρών. Όχι, περνάμε στην ακρόαση ε, του προτινόμενου Ευρωπαίου συντονιστή. Να πω, η τροπολογία, η καταληκτική ημερομήνη για την κατάσταση τροπολογιών είναι η 20 Απριλίου 12 η ώρα.